Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Ας προχωρήσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να συναντηθούμε πριν τα Χριστούγεννα. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την ημέρησα διάταξη πρώτα πρέπει να την εγκρίνουμε και βεβαίως ε, τις αποφάσεις των συντονιστών Υπάρχει και ένα σημείο για τις πράξεις καταξιοδότηση και τις ε, πράξεις εφαρμογής. Ας μην ε, καθυστερήσουμε εδώ. έχουμε βεβαίως και τη διαδικασία ψηφοφορίας εξ αποστάσεως. Ε, γνωρίζετε πλέον, είστε, είστε εξοικειωμένοι, το έχετε κάνει αρκετές φορές, δεν χρειάζεται να σας διαβάσω την όλη διαδικασία για άλλη μια φορά. Φαντάζομαι ότι δεν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα στη διαδικασία αυτή την έκτακτη διαδικασία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας υπό αυτές τις συνθήκες. Ψηφοφορία δηλαδή εξ αποστάσεως. Πρόκειται για την ετήσια έκθεση εξωτερικών σχέσεων για τα έτη 2018-2019 της συναδέλφου Κλέρ Ντέιλι. Εντάξει, εγκρίνεται η μέρη διάταξη βέβαια. Τα σημεία 4 και 14 μετατέθηκαν στην επόμενη συνεδρίαση. Το σημείο 6, εφόσον δεν υπάρχει πλέον αίτημα, απεσύρθη μάλλον το αίτημα του ECR σε ό,τι βάζει τις τελευταίε δημοκρατικέ επιθέσεις στην Αυστρία και τη Γαλλία, είχε ακυρωθεί οπότε το σχετικό σημείο. λοιπόν τις εφαρμοστικές πράξεις και την εξοδότηση πράξης τις προσπερνώ και πάμε στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως με τις τροπολογίες την, μιλάμε για την έκθεση της Claire Daily πάντα ε, και το σημείο 5 επίσης τεχνητή νοημοσύνη ερμηνεία του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, στρατιωτικές χρήσεις, ε, ε, του κατά πόσο εμπίπτουν ε, στο πεδίο της ποινική δικαιοσύνης, του ποινικού δικαίου. Λοιπόν, τώρα αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει απαρτία για την πληροφορία, οπότε παρακαλώ να μας γνωστοποιήσετε την παρουσία σας. Δεν υπάρχει ακόμα απαρτία. Δεν είναι κανείς την αίθουσα ούτως ή άλλως, απλώς ε, πατήστε το κουμπί σας, στείλτε έτσι ένα σήμα ότι υπάρχετε, ότι είστε εκεί. Εμείς δεν σας βλέπουμε βέβαια. Να ξέρουμε τουλάχιστον ότι είστε εκεί. Έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει απαρτία. Ένα άτομο μας λείπει για την απαρτία. Λοιπόν, ωραία, τα καταφέραμε. Ευχαριστώ. Και τώρα θα περάσουμε στο πρώτο σημείο ουσίας της ημέρησης διάταξης. Σημείο 7. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αισθήματα ασφάλειας, ε, μελλοντικέ ε, εξελίξεις ε, σε ό,τι αφορά τη σχετική οδηγία του Συμβουλίου για τις τρομοκρατικέ επιθέσεις και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρώτα απ' όλα θα έχω μια παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων με την επίτροπό μα, την Ήλβα Γιώχανσον, που ασχολείται με τα αισθήματα εσωτερικών και στη συνέχεια θα έχουμε την έκθεση τη Γερμανική Προεδρία Κρίστιαν ε, Κλάου, όχι για πρώτη φορά, Γενικό Διευθυντή ε, του Ομοσπονδιακού ε, Υπουργείου Εσωτερικών τη Γερμανία, τη ε, Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση λοιπόν, μέλο που έχει και την Ευρωπαϊκή Προεδρία, βεβαίω την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση Γερμανία. Να περάσουμε λοιπόν στην κυρία Γιώχανσον. Είχαμε μια συνάντηση με εμπειρογνώμονες 22 Σεπτεμβρίου. Έγινε μια μελέτη από την, ε, το Γραφείο Πολιτικής μας. Η συνάδελφος ε, Νιώβη Μαλούρα από το ε, Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Θα ακούσουμε πρώτα την Επίτροπο Γιώχανσον. 15 λεπτά maximum είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να μιλήσει και μικρότερο χρονικό διάστημα η κυρία Γιώχανσον και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Κλάους και βεβαίως ε, θα έχουμε και την ανταλλαγή απόψεων, πρώτα οι συντονιστές και μετά τα υπόλοιπα μέλη που θέλουν να πάρουν το λόγο. Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, κυρία Γιώχανσον, είστε εκεί. Έχετε το λόγο. Σα ε, ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και χαίρομαι που θα το συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τι ε, πρόσφατε ε, βίε τρομοκρατικέ επιθέσει στο Παρίσι, την Νίκαια τη Βιέννη. Πρόκειται για μια επίθεση κατά των ελευθεριών μας. Είναι επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κοινών μας έργων. Ό,τι αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελευθερία έκφρασης και πληροφορίας, πληροφόρησης, το, το δικαίωμα στην ε, παιδεία, το δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης, της ελεύθερης έκφρασης και πάνω απ' όλα το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην αγάπη. Αυτά όλα κατοχυρώνονται στον χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν και να δείξουμε ισχυρή αλληλεγγύη ω Ένωση. Θα πρέπει να ενωθούμε ως ε, κοινωνία, θα πρέπει να καταδείξουμε ότι οι αξίες μας είναι αναπαλωτρίωτες και δεν μπορούμε να αντιχαστούμε από αυτού. Είμαστε λοιπόν όλοι μαζί η Ευρωπαϊκή Ένωση και για μένα είναι σαφές ότι θα πρέπει να εντείνουμε την καταπολέμησή μας από κοινού κατά της τρομοκρατίας online αλλά και στον πραγματικό κόσμο για να προλαμβάνουμε, να προστατεύουμε, να ανταποκρινόμαστε. Και προβλέπεται λοιπόν ένα κοινό πλαίσιο για τις δράσεις μας. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας φυσικά δεν είναι κατά οποιασδήποτε συγκεκριμένης θρησκείας ή πολιτικής πεποίθησης. Κατευθύνεται κατά των βίαιων εξτρεμιστών του φαινομένου αυτού σε όλες τις εκφάνσεις, κατά των τρομοκρατών. Όλοι γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε αναλάβει πολλέ δράσει για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία σε όλε τι μορφέ. Πολλέ δράσει για να ενισχύσουμε την προστασία των ιστορικών συνόρων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Είμαστε πολύ καλύτερα προστατευμένοι σήμερα σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πολλέ αποφάσει οι οποίε δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί όπω πρέπει και θα πρέπει να εντείνουμε κατεπηγόντω και τη σκέλος τη υλοποίηση αλλά και τα κενά που υπάρχουν για την πιο στενή συνεργασία στην ασφάλεια. Θα βάλω λοιπόν, έχουμε βάλει το θέμα αυτό στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας στις 9 Δεκεμβρίου. Θα προτείνουμε λοιπόν νέους τρόπους αντιμετώπισης της τρομοκρατίας τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες εβδομάδες ήδη θα λεφθούν κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά το σκέλος της πρόληψης. Συνεργαζόμαστε με το δίκτυο και ευαισθητοποίηση για θέματα ριζοσπαστικοποίηση για να εντοπίζουμε τέτοια σημάδια εγκαίρω και να υπάρχει σωστή αντίδραση σε παράδειγμα σε ό,τι αφορά του τους καταδικασμένους φυλακή και σε ό,τι αφορά τα άτομα που βγαίνουν από τη φυλακή. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί η προστασία των κοινών χώρων. Θα πρέπει να προωθήσουμε το θέμα της ασφάλειας από τη φάση του σχεδιασμού. Ξέρουμε ότι για παράδειγμα, μια καλή πόρτα ή μια καλή κλειδαριά μπορεί να κάνει την διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Επίσης, διευθυντική συνεργασία μεταξύ των Δήμων και των κοινοτήτων, απαραίτητη στο μέλλον. σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση επιπλέον πόρων για την προστασία επίσης των πολιτών και την προστασία των κοινών χώρων μεταξύ των οποίων και η χώροι λατρείας. Επίσης, οι κρίσιμες υποδομές εξακολουθούν να ε, αποτελούν ενδεχομένω στόχους δημοκρατικών επιθέσεων. Θα προτείνουμε λοιπόν νομοθεσία μέσα στο έτος για την προστασία τέτοιων κρίσιμων υποδομών. Η επίθεση στην Βιέννη χρησιμοποίησε ένα ε, όπλο AK-47. Θα πρέπει να θέσουμε λοιπόν την ε, λαθρεμπορία όπλων στο επίκεντρο. Πολλές σχετικές ε, κράτη-μέλη δεν έχουν υλοποιήσει τη σχετική οδηγία σε ό,τι αφορά την παράνομη χρήση όπλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τονίσει αυτά στο επόμενο χρόνο σε ό,τι αφορά δηλαδή το πώς έχει υλοποιηθεί αυτή η νομοθεσία και δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε λήψη μέτρων. Τον Ιούλιο φέτος, σε μια ημέρα δράσης μόνο, καταφέραμε να βρούμε χιλιάδες ιστοσελίδες στο ίντερνετ με τρομοκρατικές οργανώσεις που έδιναν, για παράδειγμα, οδηγίες για το πώς να συνταρμολογηθεί ένα όπλο. Πολλοί σχεδίαζαν επιθέσεις. Αυτό τονίζει, θεωρώ, την ανάγκη και την κατεπίδωτο χαρακτήρα για να υλοποιηθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διάδοση τρομοκρατικού υλικού. Ελπίζω πριν τα Χριστούγεννα να μπορέσουμε να, να ολοκληρώσουμε τον τρομερή διάλογο για το τρομοκρατικό περιεχόμενο online. Οι πρόσφατες επιθέσεις κατέδειξαν εκ νέου ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει διαρρομένη και πιο εντατική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδο και θα ήθελα να τονίσω το ρόλο τη Europol για να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τι σχετικέ έρευνε. Επίσης, η αστυνομία θα πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να τσεκάρει σε ένα κοινό σύστημα, σε μια κοινή βάση δεδομένων ε, τα στοιχεία των υπόπτων, μεταξύ των οποίων και το σύστημα αιτίας. Μέχρι το 2023, λοιπόν, βασικός στόχος θα είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων αυτών, γιατί είμαστε ισχυροί όσο ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής μας. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν μεγαλύτερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ε, ζητημάτων διαλειτουργικότητας. Αυτό σημαίνει επίσης να μπαίνουν πληροφορίες στο σύστημα πληροφόρησης Schengen σε ό,τι αφορά τα άτομα τα οποία έχουν εντοπιστεί σε εθνικό επίπεδο ως ύποπτα για τρομοκρατία, για βίαιο εξτρομισμό. Όλοι αυτοί λοιπόν που μπαίνουν και βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει συστηματικά να ελέγχονται σε αυτή την βασική βάση δεδομένων προκειμένου να εντοπίζονται όλα τα άτομα στα οποία υπάρχει, για τα οποία υπάρχει επισήμανση ως αλλοδαπή μαχητές. Πέρσι, μία έκθεση της Frontex κατέδειξε ότι 22% όλων των επιβατών που περνούσαν τα εξωτερικά σύνορα δεν ελέγχθησαν Βάση του συστήματος πληροφόρηση Σέγγεν. Και αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι αποτελεί ένα σημαντικό χάσμα στην ασφάλεια, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Η ανάλυση λοιπόν τέτοιων δεδομένων είναι ένα βασικό εργαλείο για να εντοπιστούν οι γνωστοί αλλά και μη γνωστοί υποπτοί. Και είναι σημαντικό να υλοποιηθεί πλήρω αυτή η οδηγία για τους επιβάτες. Σήμερα θα συζητήσουμε συγκεκριμένα τη σημασία των εργαλείων που παίζουν το βασικό ε, ρόλο για το API και την αναθεώρηση των εργαλείων αυτών. Έχουμε διάφορα εργαλεία, διάφορα συστήματα πληροφόρησης τα οποία έχουμε υπόψη μας. Για να σας ε, διευκρινίσω λοιπόν πώς συνδέονται το Schengen, το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Schengen. Είναι ένα βασικό σύστημα όπου διάφορα άτομα με τα οποία υπάρχει επισήμανση, όπως για παράδειγμα λαδαπή μαχητές ή άλλα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Μπορεί απλά να πρόκειται για άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όχι ότι τα οποία θα πρέπει να συλληφθούν απαραίτητα. Εκεί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι συνοριοφυλακέ, το PR, πληροφορίε για ένα άτομο το οποίο πρόκειται να ταξιδέψει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όνομα, πτήση, θέση, ε, στοιχεία επιστοτική κάρτα ε, με το οποίο χρησιμοποιήθηκε να, για να αγοράσει το εισιτήριο. Αυτέ οι πληροφορίε λοιπόν αποστέλλονται. από τις αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα, προς το κράτος μέλος υποδοχής εκ των προτέρων πριν από την άφηξη του ατόμου. Το API. Είναι πολύ πιο παλιό από το PNR το σύστημα. Αυτή η οδηγία είναι του 2004. Πραγματικά πλέον παλιά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που βάζουμε με το διαβατήριό μας όταν κάνουμε στο αεροδρόμιο. Και αυτό υποδηλώνει στο κράτος υποδοχής το πότε ουσιαστικά θα γίνει η άφηξη και το ταξίδι. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, το χρειάζεται να δείχνουμε τα στοιχεία αυτά όταν βγαίνουμε από το αεροπλάνο. Το API λοιπόν περιλαμβάνει λιγότερες πληροφορίες από το PNR σήμερα, αλλά αποτελεί ένα συμπλήρωμα προς το PNR, γιατί περιλαμβάνονται εκεί τα άτομα τα οποία πραγματικά επιβαίνουν στο αεροπλάνο και πληροφορίες για την ταυτότητά τους σε ό,τι αφορά τα στοιχεία διαβατηρίου του, για παράδειγμα. Το API, όπως σας είπα, είναι το 2004 η οδηγία αυτή. Είναι παλιά. Είναι παλιά, όπω και να το κάνουμε. Η Επιτροπή προσφάτως ξεκίνησε αναθεώρηση της οδηγίας API και τα συμπεράσματά μας συνάδουν με αυτά που συμπέρανε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το API. Η συλλογή λοιπόν των δεδομένων API εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο στοιχειοδού σημασία. Αυτό το, ε, το τονίζει και η έκκληση του ΟΗΕ να χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύ τα στοιχεία API για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματο. Και επίσης ε, καταδεικνύεται αυτό από την ε, διευθυντική συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης. Επίσης, τονίζουμε μία σειρά κενών που υπάρχουν που μειώνουν την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της οδηγίας API στην πράξη. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει τυποποίηση, δεν υπάρχει εναρμόνιση επαρκώς, δεν υπάρχουν ε, αρκετά δεδομένα για τις δικλείδες ασφαλείας. Δεν υπάρχει επίσης συμμόρφωση με τις τελευταίες πολιτικές και ε, τις νομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αντιμετωπιστούν λοιπόν αυτά τα προβλήματα, ξεκίνησε μια μελέτη δικτύπου σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του χρόνου θα γίνει μια αναφορική πρόταση για να τροποποιηθεί, να, να ανθεωρηθεί η οδηγία API. Τι κοιτάμε, τι εξετάζουμε. Καταρχάς, να βασιστούμε στο σύστημα αιτίας για να υπάρξει streamlining των ε, δεδομένων σε οικονομίες κλίματος. Κατά δεύτερον, με τις νέες τεχνολογικές λύσεις να αυξήσουμε την ποιότητα των δεδομένων. Για παράδειγμα, να αντικατασταθεί η χειροκίνητη καταχώρηση με αυτόματη συλλογή των στοιχείων API. Για παράδειγμα, μέσω σκαναρίσματος των ε, διαβατηρίων, να μην περνούνται όλο με το χέρι. Κατά τρίτον, να υπάρξει μεγαλύτερη συλλογή δεδομένων και σε άλλες οδούς και τρόπους μεταφορών. Η τρέχουσα οδηγία δεν διευκρινίζει για ποια πτήση θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα. Αυτό επαφείται στα κρατημέλη. Αυτό που διευκρινίζει είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι συλλογή στοιχείων για εισερχόμενες πτήσεις που μπαίνουν στο Σέγγεν δηλαδή. Μία αναθεωρημένη οδηγία ενδεχομένως να καλύπτει όλες τις οδηγίες, για παράδειγμα και πτήσεις μεταξύ των χωρών Σέγγεν ή θα κάλυπτε ενδεχομένως και άλλες ε, εταιρείε μεταφορών ε, μέσω του δρόμου, για παράδειγμα. Κατά τρίτον, δεκατάρτον μάλλον, εναρμόνιση με τα στοιχεία της οδηγίας PNR. Στη φάση αυτή εξετάζουμε ενδεχόμενες λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία API με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι σημαντικό λοιπόν να τα κοιτάξουμε όλα αυτά με ανοιχτό πνεύμα, να ανταλλάξουμε απόψει για όλα αυτά τα θέματα. Και προσβλέπω στην διαδικασία αυτή. Το πριν δεν είναι μία βασική δάση δεδομένων, ούτε περιλαμβάνει στοιχειώδη δεδομένα. Είναι μία βάση δεδομένων ποινική απόφαση επικρίνουμε επίσης είναι επίσης παλιά, του 2008. Και μας επιτρέπει συλλογή DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων, hit no hit και στοιχεία καταχώρησης. Μόνο τα άτομα ή τα οχήματα τα οποία αποτελούν τμήμα ποινική έρευνα συμπεριλαμβάνονται στην βάση δεδομένων αυτών. Οι εθνικές αρχές λοιπόν μπορούν να στραφούν σε εθνικές αρχές άλλων κρατών μελών και να λάβουν διμερείς ανταλλαγή στοιχείων. Το πρίμι, λοιπόν ουσιαστικά αποτελεί ένα σύνδεσμο για να δούμε κατά πόσον υπάρχει επισήμανση σε σύστημα άλλου κράτους μέλους. Αν λοιπόν η αστυνομία ενός κράτους μέλους έχει δακτυλικά αποτυπώματα σε μια ποινική έρευνα από ένα έγκλημα, και δεν ξέρουν σε ποιον ανήκουν τα, κάτι, τα δακτυλικά αποτυπώματα αυτά, τσεκάρουν στην εθνική βάση δεδομένων και δεν βρίσκουν αντιστοιχεία των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πριν για να υπάρξει σύγκριση με τα συστήματα άλλων κρατών μελών και αν υπάρχει αντιστοιχεία μπορούν να στραφούν στα κράτη-μέλη αυτά για να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων και στα στοιχεία αυτά τα οποία χρειάζονται. Αυτή η έλεγχη είναι βασική στι ποινικέ ερευνέ και μα βοηθούν να εντοπίσουμε πολλού εγκληματίε. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις έρευνε αυτές μόνο βάσει εθνικών ε, βάσεων δεδομένων. Όταν ελέγχουμε λοιπόν δακτυλικά αποτυπώματα, μπορούμε να δούμε για παράδειγμα ότι δεν υπάρχει ολικό δακτυλικό αποτύπωμα, είναι μονομερικό. Αλλά μπορεί να υπάρχει σύγκριση μέσω του συστήματο για να βρεθεί το συνολικό τελικά δακτυλικό αποτύπωμα. Και έτσι ενδεχομένω προβαίνουμε σε αναγνώριση και εντοπισμό των υπόπτων και οδηγούμαστε σε δίωξη και καταδικάση των ε, υπετίων. Είναι παλιά η νομοθεσία αυτή όμω, από το 2008. Από τότε καταλαβαίνετε ότι η τεχνολογία, το περιβάλλον, ε, ε, όλα έχουν εξελιχθεί και αλλάξει. Και η λειτουργικότητα των συστημάτων, το privacy by design, οι τεχνικές λύσεις, η έγκριση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου το 2016. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση πριν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε μια έκθεση εφικτότητας για την βελτίωση της απόφασης πριν το Μάιο φέτος. Αυτή η έρευνα λοιπόν και η έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την οποία ζητήσατε πριν από δύο χρόνια και άλλες αναλύσεις που έχουν γίνει από άλλους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και σχετικές συζητήσεις που έχουν γίνει για το πριν στο Συμβούλιο έχουν καταδείξει τις βασικές ελλείψεις που υπάρχουν στο σύστημα πριν και τόνισαν και ενδεχόμενες ε, λύσεις. Πρέπει καταρχάς να απλοποιηθεί το πριν. Έχουμε 351 συνδέσμους μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρχουν κατηγορίες δεδομένων. Ένα κράτος μέλος, για παράδειγμα, ψάχνει δεκλικά αποτυπώματα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει στην φάση αυτή να πάει σε κάθε κράτος μέλος να τσεκάρει κατά πόσον υπάρχει δυστυχία. Αν θέλει να ψάξει DNA, αντιστοιχεία DNA, θα πρέπει να μεταβεί σε άλλο κανάλι για να δει κατά πόσον υπάρχει αντιστοιχεία. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν υλοποιήσει την απόφαση πριν. Μπορεί να υπήρχε, για παράδειγμα, αυτού ένα κεντρικό ρούτερ για τον σύνδεσμο αυτό. Αυτό θα διευκόλυνε πάρα πολύ την συνδέσεις μεταξύ κρατών μελών. Ένα κεντρικό ρούτερ λοιπόν θα είχε και άλλα πλανεκτήματα συλλογή στατιστικών στοιχείων, τεχνική αρρωγή και αυτό σημαίνει ότι ένα κράτο μέλος θα μπορούσε να μπει σε ένα σύνδεσμο και να ελέγξει η αντιστοιχεία των στοιχείων αυτών σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν έχουμε κατά νου, να απλοποιήσουμε τη ροή των πληροφοριών με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι ένα κεντρικό ψήφι των πληροφοριών πριν, έτσι. Όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα βασίζονται στα κράτη-μέλη δεν έχουν τα άλλα κρατημέλη άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των άλλων. Και βεβαίως υπάρχει, τα λειτουργεί το σύστημα hit no hit. Πρέπει βεβαίω να επιταχύνουμε και να ευθυγραμμίσουμε την αλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, εμπειρογνωμόνων σε ό,τι αφορά τα επιβεβαιωμένα hit. Σε ό,τι αφορά ε, τα ανώνυμα hit τώρα ε, και τα δακτυλικά αποτυπώματα, ε, δεν χρησιμεύει αυτό μια ποινική δίωξη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, να ταυτοποιήσουμε τον άνθρωπο. Τον... Συγγνώμη, ε, λέει ο Πρόεδρος, σας είχαμε δώσει 15 λεπτά και μιλάτε ήδη 19, οπότε ε, σας παρακαλώ, διότι πρέπει να ακούσουμε και τη Γερμανική Προεδρία, τους συντονιστές, τους ομιλητές. Ναι, θα πρέπει να επιταχύνουμε τις αποφάσεις πριν, έτσι ώστε να υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία ευθυγράμμιση της αλλαγής δεδομένων και αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τη μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά το πριν. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ κυρία Γιώχανσον ε, που ολοκληρώσατε την παρουσίασή σας έτσι ώστε να ακούσουμε και τον Δόκτωρ Κλώσ και στη συνέχεια βεβαίως να δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους. Είχετε πέντε λεπτά κύριε Κλός. Ναι, εδώ είμαι, δεν ξέρω αν με βλέπετε. Όχι, δεν σας βλέπουμε. Ελπίζω να μην έχουμε κάποια δυσκολία. Πέντε λεπτά, Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν σας βλέπουμε ακόμα, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, τώρα σας βλέπουμε. Επιτέλους. Και με ακούτε κιόλας. Ναι. Έχετε το λόγο. Για πέντε λεπτά. Πολύ ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ και που μου δίνετε την ευκαιρία. Είχα την ευκαιρία και την προηγούμενη εβδομάδα να κάνω παρουσίαση. Πάλι όμως χάσαμε Α. Υπήρξε η κοινή δήλωση του Συμβουλίου, των Υπουργών Εσωτερικών, της περασμένης Παρασκευής. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ όλος ιδιαίτερος σε αυτή την κοινή δήλωση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης αλλά και αποφασιστικότητας για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Και βεβαίως το πιο σημαντικό στοιχείο, πιστεύω, είναι η δομή της κοινή δήλωσης. Δεν αναφερόμαστε εκεί μόνο στα κλασικά ζητήματα της ασφάλειας. Λέμε ότι εδώ υπάρχει ένα πλαίσιο πολύ ευρύτερο και χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα οι Υπουργοί επανεπιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Δεν ξεκινάμε δηλαδή από το μηδέν. Προσαρμοζόμαστε διαρκώς απέναντι στην απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας. Και βεβαίως και μας επηρέασαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις και στις εργασίες μας. Έχουμε λοιπόν και ένα σχέδιο συμπερασμάτων για την εσωτερική ασφάλεια και πολλά από τα σημεία δράσης θα τα βρείτε σε αυτό το έγγραφο της Γερμανικής Προεδρίας που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Υπουργών του Δεκεμβρίου Πάντως σε αυτή την κοινή δήλωση το πρώτο που αναφέρουμε είναι η αρχή της θρησκευτική ελευθερίας. Δηλαδή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν στρέφεται κατά κάποιων θρησκευτικών πεπιθήσεων. Είμαστε κατά του ακραίου βίαιου εξτρεμισμού. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η σφαιρική προσέγγιση και βεβαίω υπάρχει υπάρχουν και τα ζητήματα τη κοινωνική συνοχή και τα μέτρα κοινωνική συνοχή που πρέπει να παρθούν. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτή την αίσθηση του ανήκειν στις κοινωνίε μας. Και αυτό έχει να κάνει με την ενσωμάτωση, με την ένταξη. Οι υπουργοί είπαν ότι βεβαίως αυτό ε, έχει δύο όψεις. Πρέπει ο ίδιος ο πρόσφυγας, ο μετανάστης να συνεισφέρει στην ένταξή του, την, την επιτυχή ένταξή του, αλλά και οι αρχές, οι θεσμοί της χώρας υποδοχής ε, να του παράσχουν το κατάλληλο πλαίσιο. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στα ζητήματα ασφάλειας, βεβαίως το θέμα του χώρου Σέγγεν, τη σημασία του να θωρακίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα, δίνοντας βεβαίως έμφαση εδώ ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόληψη ε, σε ό,τι αφορά την, εισόδου, την είσοδο μάλλον ε, ανθρώπων που αποτελούν απειλή για τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν ε, μια μεγάλη πρόκληση για τις δυνάμεις ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να σημειώσουμε να μπορούμε να παρακολουθούμε την κινητικότητα, της κινήσεις αυτών των ανθρώπων και εκεί έχει σημασία η βελτίωση της ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Αυτό συνδέεται και με την ε, ε, σύμπραξη, αν θέλετε, τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών, να μπορούν δηλαδή οι αστυνομικέ αρχέ κάθε χώρα να έχουν πρόσβαση στι πληροφορίε που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά του και να χρησιμοποιήσουμε βεβαίω ε, και τι ήδη υπάρχουσε γνώσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μια ανταλλαγή πληροφοριών πληροφοριών που υπάρχουν ήδη, αλλά όπω είπαν οι υπουργοί είναι σημαντικό να, η συλλογή δεδομένων, η ανάλυση δεδομένων, η διάδοση των δεδομένων αυτών, σεβόμενοι πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έγινε και μία αναφορά στην κοινή δήλωση 21 Οκτωβρίου ε, για το μέλλον τη. Europol, μια και η Europol παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ε, με το, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας, και ένα άλλο ζήτημα είναι η πρόληψη της ε, και επιγραμμικά και στο διαδίκτυο και έγινε αναφορά στις, ε, στο σχετικό κείμενο στον κανονισμό για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο θέλουμε να ακολουθεί μια γρήγορη διαδικασία εδώ είναι, υπήρξε ένα σαφές μήνυμα από πολλούς υπουργούς, πολλούς υπουργούς ε, στις παρεμβάσεις τους ότι ε, ελπίζουν ότι θα ολοκληρώσουμε το φάκελο αυτό και θα μπορέσει αυτή η σημαντική νομοθεσία να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αναφέρθηκε και την περασμένη Δευτέρα, είναι το θέμα της κρυπτογράφησης των στοιχείων και τη δυνατότητα που θα έχουν οι αρχές επιβολής του νόμου με μια συγκεκριμένη διαδικασία screening να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ένα άλλο στοιχείο που έχει σημασία είναι η ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών για αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούν απειλή, τρομοκρατική απειλή, το θέμα των ξένων μαχητών και βεβαίως ε, έγινε αναφορά στα μίντια για το πόσο πρέπει να ορίσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να έχουμε ένα κοινό ορισμό. Δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι τι καταλαβαίνει το κάθε κράτος μέλος ως απειλή για το έδαφος του. Και αυτό αρκεί για να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει τα 5 λεπτά, Πρόεδρε. Θα ήθελα όμως να πω, διότι είναι το ζήτημα κλειδί αυτό είναι η δομή, η αρχιτεκτονική της ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε μια φορά στην πρωτοβουλία API, την οποία προφανώς υποστηρίζουμε, αλλά και θεώρηση του συστήματος PRIM. Είπε πολύ καλά η Επίτροπος, ε, το ανέφερε πολύ καλά το πώς πρέπει να τροποποιηθεί αυτό. Συγγνώμη, ε, ε, για την καθυστέρηση. Είχαμε ένα πρόβλημα με την κάμερα στην αρχή, γι' αυτό είμαι έτοιμο πάντω να απαντήσω στα ερωτήματά σα. Sure Ευχαριστούμε, δόκτωρα Κλώσο. Θα παρατηρήσατε ότι έχουμε προβλήματα γιατί η κάμερα σας έχανε όλη την ώρα. Οι διερμηνείς, τους οποίους ευχαριστούμε, συνέχισαν παρά το γεγον τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες δυστυχώς αποτελούν καθημερινότητα πλέον στη δουλειά μας. Αλλά ας προχωρήσουμε τώρα στον ανοιχτό διάλογο που θα μας απασχολήσει αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταρχάς ένα πρώτο γύρο ομιλητών, τους συντονιστές, για το, τους ονόματος του ΕΛΚ, κύριος Μάντελ πρώτα. Αν είστε εκεί παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σας Επιτροπέ να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Γερμανικής Προεδρίας για τις ε, χρήσιμες πληροφορίες. Θα ήθελα ως Αυστριακός να σας εκφράσω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα συλλεπιτήρια και την πρακτική υποστήριξη η οποία ήλθε από όλες τις πλευρές της Ευρώπης μετά από τις φρεχθές και βίαιες αυτές επιθέσεις στη Βιέννη δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρώτη επίθεση που έλαβε χώρα στην Ευρώπη και θα πρέπει όλοι να εργαστούμε σκληρά να είναι, αν όχι η τελευταία αυτή η επίθεση, εν πάση περιπτώσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να μην έχουν έφορο οι τρομοκράτες στην Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει να αλλάξει και η ιδεολογία του πολιτικού Ισλάμ. Γιατί δεν είναι μόνο οι τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και η πολιτική ιδεολογία του πολιτικού Ισλάμ και φυσικά και ό,τι αφορά τους εκπροσώπους του πολιτικού Ισλάμ. Γι' αυτό υποστηρίξω, υποστηρίζω όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτρεπός για το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών που έχει κενά και θα πρέπει να καλυφθούν αυτά τα κενά. Σε ό,τι αφορά και τους ανθρώπους εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούν το πολιτικό Ισλάμ από τη Συρία και από άλλα μέρη. Ξέρουμε ότι άνθρωποι έρχονται από εκεί στην Ευρώπη και θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών να τα καλύψουμε με όσο λιγότερη γραφειοκρατία γίνεται και όσο πιο εκτενώς γίνεται για να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να αποτελέσουν και τμήμα του νέου πακέτου ασύλου του Δεκεμβρίου και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διάδοση διαλογών, ιδεολογιών μίσους online και offline αυτού του πολιτικού Ισλάμ. Αυτό προφανώς και αποτελεί καθήκον και δουλειά κρατικών φορέων. Δεν μπορούν να τα αναλάβουν αυτό μόνο οι ιδιώτες. Φυσικά οι ιδιώτες πρέπει να συμβάλλουν σε ό,τι αφορά την υποδάφλεση μίσους, όλα αυτά δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα. Ούτε μπορεί να υπάρχει ατιμορρησία για τέτοιου είδους υποδάβληση μίσους και τέτοια επικίνδυνα περιεχόμενα. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε εντατικά για τέτοια θέματα και μάλιστα με ποιοτικά αποτελέσματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από κοινού όλους αυτούς που θέλουν να μας αποδυναμώσουν από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους αυτούς που θέλουν να διχάσουν την κοινωνία μας και θέλουν να μας φέρουν αντιμέτωπους μεταξύ μας. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Θα πρέπει να εργαστούμε συνεκτικά από την πολιτική ιδεολογία μέχρι την καταπολέμηση του πολιτικού Ισλάμ. Ο πρόεδρος διακόπτη, κύριε Λούκασε και ας ε, προωθήσουμε, λέει ο κ. Λούκας, και κοινοβουλευτικά αυτό το έργο. Κύριε Λούκα, παρακαλώ, μην ξεχνάτε ότι έχετε δύο λεπτά ο κάθε συντονιστή. Οπότε παρακαλώ να το τηρείτε, είμαστε αυστηροί. Έχουμε λίγο χρόνο τη σήμερα ημέρα και πρέπει διαρκώς να έχουμε στο μυαλό μας το χρόνο. Έχετε το λοιπόν υπόψη συνέχεια, τελείω ξεφεύγει η κατάσταση. Και τώρα έχει το λόγο η Κατερίνα Κινίτσι. Παρακαλώ, προσπάθησε Προσπαθήστε να εκφραστείτε σύντομα. Δύο λεπτά. Κατερίνα, έχετε το λόγο. Χωρίς εικόνα η ομιλήτρια. Eh, voglio ringraziare in particolare la commissaria Johansson per aver sottolineato e aver preannunciato la nuova agenda per la lotta al terrorismo. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και το επιτελείο της για την ανταλλαγή ε, πληροφοριών για την ενημέρωση και για τη βελτίωση της δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Η Κομισιόν έχει προβλέψει την ε, ε, ενημέρωση της οδηγίας API, Advanced Passenger Information. Ε, αυτή η ενημέρωση, εξυγχρονισμός χρειάζεται. Μπορείτε να μας δώσετε όμως και κάποιες ημερομηνίε για πότε δηλαδή μπορούμε να περιμένουμε σχετική ε, ε, ημερομηνία. Έπειτα, για τις αποφάσεις ΠΡΟΜ, Και γι' αυτό είπατε πως είναι πια ξεπερασμένο, πεπερασμένο σύστημα. Θα έπρεπε λοιπόν να εξυγχρονιστεί και από τεχνικής άποψης. Και θέλω να σας κάνω την εξή ερώτηση. Οι αποφάσεις ΠΡΟΜ, όπως και άλλα μέσα αστυνομικής συνεργασίας, χρησιμοποιούνται στις ε, τρομοκρατικές ε, ε, και σήμερα ακόμα είπατε πω υπάρχουν ελλείψεις στη μεταγραφή αυτών των αποφάσεων όσον αφορά την τρομοκρατία όπως αυτή ορίζεται στη σχετική οδηγία. Εάν πρέπει, μάλλον σκοπεύετε να παρέμβετε ως Κομισιόν και για αυτή την πτυχή και πώς. Και ακόμα μια ερώτηση για την Europol. Όπως γνωρίζουμε, η Europol ε, παίζει κεντρικό ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών και γνωρίζουμε πως θα πρέπει να ε, ε, σύντομα να ασχοληθούμε με την νέα εντολή της Europol. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν την Επίτροπο αν μπορεί να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες, περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα καταφέρουμε να καταστήσουμε την συνεργασία της αστυνομίας, όχι πλέον ad hoc, δηλαδή ένα περίπτωση και περιστασιακά, αλλά ουσιαστική, μόνιμη και διαρκή. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την προσήλωσή σας στο θέμα της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Ευχαριστώ ειλικρινά. Και εμείς ευχαριστούμε η Φαμπιέν Κελέρ τώρα για δύο ε, λεπτά. Φαμπιέν. On peut peut pas vous écouter.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 Fabienne, ça ne vous dérange pas αν δεν σα πειράζει θα δώσουμε το λόγο στον Patrick ε, των Πρασίνων. Σα παρακαλώ να ετοιμαστείτε το μεταξύ εσείς για να πάρετε το λόγο. Πάτρικ, εσύ είσαι εκεί. Ναι, έτοιμος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την τραγωδία των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθήσεων, θα, τον, θα ήθελα να πω ότι όλοι έχουμε σοκαριστεί με το τι έγινε. Ποτέ δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε τι αξίε μα, αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία λόγου, που, α, ε, όπως ας πούμε ο Σαμουέλ Λαμπατή ακριβώς γι' αυτό πέθανε, γι' αυτό σκοτώθηκε. Ε, θα πρέπει ε, να μην αυτοπεριορίζουμε τις αντιδράσεις μας αυτές σε μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις. Τώρα η αστυνομία ε, έχει αποτύχει να παρακολουθήσει τους δράστες, όπως ε, ας πούμε στην περίπτωση του, του δράστη της Αυστρίας, ε, ενώ ήταν σε σημασμένη Επίτροπε, δεν υπάρχει ε, πιστεύω έλλειψη ε, στις ε, αρμοδιότητες επιβολής αλλά στην επιβολή την ίδια. Εσείς συμφωνείτε και έπειτα. λείπει το στοιχείο της ε, αναφοράς από την πρότασή σας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πώς οι τρομοκρατικές ενέργειες όντως θα διώκονται. Θα ήθελα να γνωρίζω επίσης πώς ε, ε, θα διαδοθεί η συλλογή πληροφοριών μη υπόπτων ταξιδιωτών στην Ένωση, πληροφορίες δηλαδή επιβατών για ταξίδια με τρένο ή με ferry boat δεν έχουμε πλέον δηλαδή δυνατότητα να ταξιδεύουμε ανωνύμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κομμάτι της ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ένωσης. Γνωρίζετε πως το Συμβούλιο δεν υιοθέτησε το ψήφισμα της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του PNR, γιατί ακριβώς είναι ιδιαίτερα επίμαχο το ζήτημα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τώρα έχει εγγύψει στην μελέτη της οδηγίας PNR. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι είναι δυσανάλογο να κρατώνται στοιχεία των επιβατών για χρόνια. Μπορώ να σας ρωτήσω πότε θα υποβάλλετε πρόταση για να της οδηγίας οδηγίες ώστε αυτή να καταστεί συμβατή με τα θεμελιώδη δικαιώματα και Επίσης, θα αρχίσετε διαδικασία κατά παράβαση για τα κράτη που δεν συμμορφώνονται με τις τελευταίες σχετικές αποφάσεις στο δικαστήριο και μια τελευταία παρατήρηση για την κρυπτογράφηση. Έχουμε συζητήσει ξανά το θέμα, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ασφάλεια και πρέπει να αποφασίσουμε ανάμεσα στις ασφαλείς επικοινωνίες και την δυνατότητα ε, κάλυψης ή ανακάλυψης ε, θα είστε έτοιμοι να καταστήσετε την κρυπτογράφηση λιγότερο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Τώρα, Φαμπιέν Κέλλερ, είστε έτοιμοι. Είναι πάλι η σειρά σας. Έχετε το λόγο εάν είστε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε λέει η κυρία Κέλλερ. Ε, συγγνώμη για την δυσκολία αυτή την τεχνική. Κυρία Πίτροπη, κύριε Γενική Διευθυντή, ευχαριστώ πολύ για την απόλυτη σας αφοσίωση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την υπεράσπιση των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ κύριε Κλώση για τη συγκεκριμένη σας δουλειά, για την κλείσιμο του ντοσιέ, για την ε, γραφή τρομοκρατικού περιεχομένου online. Ε, ε, εσείς κάνατε προσπάθειες για βελτίωση της οδηγίας αλλά και ε, για βελτίωση των, των αποφάσεων προύμα. Μπορείτε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα για το πώς θα εξασφαλίσουμε την καλύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ε, πληροφοριών των κρατών μελών και εάν προβλέπετε τη δυνατότητα να συνδέσετε το σύστημα ή τη συμφωνία ΠΡΟΥΜ με τους διαχειριστές των βάσεων δεδομένων ε, και δεύτερη ερώτηση και για τους δύο για ένα άλλο θέμα που είναι το Brexit. Πιστεύετε το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει στο, στις αποφάσεις ΠΡΟΜ και να ανταλλάσσει στοιχεία δεδομένα με τα κράτη-μέλη του Ένωσης. Ξέρετε πως υπήρχε πρόβλημα στην προστασία του, ε, των δεδομένων από την Μεγάλη Βρετανία μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια η Μεγάλη Βρετανία είναι μια σπουδαία χώρα και εδώ θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία, είναι απαραίτητη η συνεργασία όσον αφορά τα θέματα τρομοκρατίας με αυτό τον μεγάλο μας γείτονα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στον κύριο Πατρίκη Τζακή από το ECR. Πιέσε το κουμπί της ομιλίας, σε παρακαλώ. Ναι, ωραία. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά. Υπάρχουν νέα στοιχεία που είναι σημαντικά. Πρώτον για τη μετανάστευση. Δεύτερον, ε, Δεύτερον είναι πού στρατολογούν οι τρομοκράτες. Ε, καταρχάς λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ε, σύστημα το οποίο να είναι καθολικό και να μπορεί να μας προστατεύσει από τις αφήξεις ανθρώπων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά και μόνο για να ε, προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Πρέπει να βρούμε αποτελεσματικά εργαλεία σε αυτό το τομέα. Δεύτερον, ποιοι, ποιες είναι οι περιοχές στρατολόγησης. Το ίντερνετ ε, πρώτα απ' όλα και ε, γι' αυτό η ερώτησή μου προς την Επίτροπο είναι πώς θα μπορέσουμε να κάποια μέρη έτσι ώστε να στηρίξουν λύσεις ε, για την καταπολέμηση του τρομοκρατίας στο ίντερνετ. Εννοώ την κανονισμό περί τρομοκρατικού περιεχομένου επιγραμμικού. Και εδώ θέλω να, τώρα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις ιδέες σας, για την συνέχιση της εργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα ε, ε, ευαίσθητη πληροφορία που μπορεί να παίξει ρόλο κλειδί σε πολλούς τομείς και να ε, προλάβει την τρομοκρατία. Θα πρέπει να καταπολεμούνται οι τρομοκράτες εκεί όπου βρίσκονται, δηλαδή στο ίντερνετ και στις και στις νέες πλατφόρμες για τη γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Αυτές τις πλατφόρμες χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γιάκη. Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Έρνστα από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Αλλά ένα πράγμα να πω. Όταν μιλάμε για τρομοκρατία, να διευκρινίσουμε τι εννοούμε, ποιον εννοούμε. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος το είπε και ο Υπουργός Ζεχόφερ ε, στη Γερμανία. Είναι ο εξτρεμισμός ο δεξιός. Να ξέρουμε τι συζητάμε. Φυσικά μιλάμε για την Ισλαμική τρομοκρατία. Αυτό είναι σαφές. Υπάρχει και αυτή η μορφή της τρομοκρατίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει διάκριση και ο δεξής ε, εξτρεμισμός είναι δύσκολος. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τι ακριβώς συζητάμε σε πρώτη φάση και να ρωτιέμαι αυτό που ακούμε, δεδομένα, δεδομένα, δεδομένα ακούμε. Αυτό μπορεί να προλάβει τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτή είναι η ερώτηση. Είπατε γιατί δεδομένα πριν ότι χρειαζόμαστε επίσης την ε, ε, οδηγία του 2004 η οποία θα πρέπει να ανανεωθεί και θα πρέπει να σας πω με πάσα ειλικρίνεια ότι ανησυχούμε. Ανησυχούμε ιδιαίτερως ότι πού θα σταματήσει η κατάσταση αυτή στα κράτη-μέλη. Η οδηγία για το DNA ήταν σαφέστατη το 2017. Τι έχει γίνει όμως και θα ήθελα να ζητήσω να μας το πει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς έγινε στην υλοποίησή της και θέλετε λοιπόν να μαζεύετε παντού δεδομένα όπου και να βρίσκεται κανείς. Στο σιδηρόδρομο, στο λεωφορείο, σε, σε κτίρια, παντού. Αυτό πιστεύετε ότι θα μας κάνει πιο ασφαλείς και εμάς και τη ζωή μας. Θέλουμε να ζητήσουμε λοιπόν κάτι παραπάνω και ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί υπάρχει τρομοκρατία αλλά θεωρώ ότι μόνο σε περιορισμένο βαθμό μπορούμε να μειώσουμε τέτοια φαινόμενα με αυτόν τον τρόπο που προτείνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τους μη εγγεγραμμένους η Λάρα Φεράρα. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις μας θύμισαν ακόμα μια φορά πόσο πολύ η τρομοκρατία είναι ε, ύπουλη, χτυπά εκεί που η προσοχή έχει λίγο αποσπαστεί και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να εφησυχαζόμαστε και κυρίως πρέπει να ποντάρουμε πάντα στην πρόληψη την νομική και την κοινωνική και σίγουρα χρειάζεται να βελτιώσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή αμέσως τη διαλειτουργικότητα των ε, ε, τραπεζών δεδομένων όπως και να υπάρξουν ε, διαθεσμική συνεργασία για τις ηλεκτρονικές, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και επίσης να μεταγραφούν αμέσως οι οδηγίες κατά του, της ανακύκλωσης βρώμικου χρήματος σε όλα τα κράτη έτσι ώστε να μπορούμε να αναχαιτήσουμε τη χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων όπως είναι και οι τρομοκρατικές. Μια ερώτησή μου προς την Επίτροπο αφορά ένα άλλο θέμα, δηλαδή την, το Σέγγεν. Αυτές τις μέρες γίνει και λόγος για τη μεταρρύθμιση του Σέγγεν επειδή δυστυχώς αναπόφευκτα όταν συμβαίνουν τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις ε, βλέπουμε τη σύνδεση πάλι μεταξύ μετανάστευσης και ε, τρομοκρατίας. Αυτή η πρόταση λοιπόν για μεταρρύθμιση του Σέγγεν που προτάθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση ε, βρίσκει σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν προχωρεί προς την κατεύθυνση αυτού που να, δου, του επανεξετάσουμε αυτού, αυτόν τον πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί γιατί αν πρέπει να ενεργήσουμε χρειάζεται να ενεργήσουμε ε, για όλες τις πτυχές που απαρίθμησε η Επίτροπε πώς από ο ρυθμιστικής άποψης. Μάλιστα, ευχαριστώ. Δεύτερος γύρος ομιλητών τώρα. Και βέβαια μετά θα επανέλθουμε στους κεντρικούς μας ομιλητές. Επίτροπε, την Επίτροπο Γιώχανσον και τον δόκτωρα Κλώσ της Γερμανικής Προεδρίας. Αλλά να τελειώσουμε πρώτα με τις ερωτήσεις γιατί έχουμε ακόμα μερικά λεπτά. Λοιπόν, από πλευρά του ΕΛΚ είναι η Ιζαμπέλ Βίσλερ Λίμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι ε, και εγώ αλλά και άλλα μέλη θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να πρεσβευτούμε τις αξίες μας. Πρέπει δηλαδή να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ ε, του καθήκοντος να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές ε, από τρομοκρατικές επιθέσεις και να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε αγαθοί, διότι οι εγκληματίες δεν είναι αγαθοί. Θα ήθελα, να, κυρία Επίτροπε, να ρωτήσω, η σχέση με το Βασίλειο ε, τι συνεργασία θα έχουμε στο μέλλον. Θα ήταν κρίμα πραγματικά να χαθεί αυτή η πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών ε, που ε, έχει στη διάθεσή της στον Ηνωμένο Βασίλειο, διάθεση του Κάτι άλλο. Θέλουμε να τελειοποιήσουμε το πριμ. Πολύ σημαντικό αυτό. Η Κομισιόν έχει όμως προβλέψει ένα χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Βεβαίως ε, εγώ ε, είμαι απολύτως πεπισμένη ότι πρέπει να συντηρήσουμε το χώρο Σέγγεν, το κοινό χώρο μας, αλλά για να τον συντηρήσουμε, να τον διατηρήσουμε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι και ασφαλής. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ισαμπέλ Σάντος τώρα, S&D. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ισαμπέλ Σάντος. Thank Mr. President. While we strongly... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς ε, βεβαίως καταδικάζουμε κάθε μορφή τρομοκρατίας, όμως είναι σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να καταλάβουμε τις ρίζες της τρομοκρατίας αυτής. Η πρόταση περί ασφάλειας ε, των Υπουργών Εσωτερικών της Περνόμενης Παρασκευή, ε, βεβαίως είναι σημαντική και αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής καταπολέμησης τρομοκρατίας. Όμως δεν μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος. Μια κοινή απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Δεν μπορούμε ε, να ε, απαρνηθούμε τις βασικές μας, τις θεμελιώδεις αξίες μας, ε, τις αρχές μας. Ε, η συζήτηση για το Σέγγεν δείχνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλες προοπτικές που μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα πιο μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Επίτροπε να σας ρωτήσω Πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το νέο σχέδιο δράσης για την ένταξη και την ενσωμάτωση και ποιος θα είναι ο ρόλος των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και των Δήμων σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ και τώρα Renew. Κυρία Μάιτερα Σατούρλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί, έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα σε επίπεδο τρομοκρατία και πρέπει να το προσαρμοστούμε κι εμεί. Κάτι που μπορούμε να υπογραμμίσουμε είναι ότι η συνδεσιμότητα μεταξύ των βάσεων δεδομένων που συμμερίζονται τα κράτη-μέλη δεν είναι ε, η καλύτερη δυνατή σε όλα τα κράτη-μέλη. Με ανησυχεί ιδιαίτερα και η νέα τάση ριζοσπαστικοποίηση, βία ριζοσπαστικοποίηση, διότι είναι πιο εύκολο μέσω του ίντερνετ να δημιουργηθούν κοινότητες μίσους. Και μέρος αυτών των κοινότητων μίσους, μπορεί στη συνέχεια να μετατραπούν σε συγκεκριμένες ομάδε ε, ομάδες κρούσης ε, που οδηγούν σε βία και σε ε, δολοφονία. Έχουμε τους νεοναζί, τους ακροαριστερούς, τους νεον, ε, Είναι πολλά τα στοιχεία που μας υποχρεώνουν να εξυγχρονιστούμε. Υπάρχει ε, μια έκθεση ε, της Europol ε, ε, στη χώρα των Βάσκων όπου μας λέει ότι το 2020 αυτή η έκθεση ότι υπάρχουν νέες απειλές δημοκρατικές. Λοιπόν, ποιες είναι οι τάσεις, οι πληροφορίες που έχουμε για διάφορες τάσεις ριζοσπαστικοποίησης στα κράτη-μέλη. Υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Βάιμερς. Είστε συνδεδεμένος κύριε Βάιμερς. Μπορεί να πατήσετε το κουμπί παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Όχι, ε. Δηλώνει ότι ενδεχομένω οι τρομοκράτε μπορεί να χρησιμοποιούν του οδού μετανάστευση. Και ο Guardian θεωρεί ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του φαινομένου αυτού. Και ότι ο άνθρωπος ο οποίος δολοφόνησε τον δάσκαλο στην Γαλλία ήταν μετανάστες. Είναι λάθος αυτή η ισχυρισμή του Guardian και σε ό,τι αφορά τι δηλώσει του Μακρόν. Υπάρχει όμω, είναι προφανέ, μία σύνδεση μεταξύ τη μετανάστευση και τη τρομοκρατία. Λέμε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Και νομίζω ότι έτσι ολοκληρώσαμε, μάλλον με άλλου τρει ομιλητέ, θα ολοκληρώσουμε τον δεύτερο γύρο. Είστε online. Nope, nope. Then how about Moritz Körner, Renew? Από το Renew. Α, ο Μπάλας Χιτζβέγγι. Ναι, με ακούτε? Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ την Επίτροπε για τα σχόλια της. Θα ήθελα να θίξω δύο θέματα. Πιο πολλά. Μάλλον είχαμε παραπάνω από δύο τρομοκρατικές επιθέσεις. Και στη μία περίπτωση ε, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Μεσογείου και μετά χάθηκαν τα ίχνη του. Και ο δεύτερος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στην Αυστρία και στράφηκε κατά των συμπολιτών του. Και στις δύο περιπτώσει καταδεικνύεται η δυσκολία της ε, ενσωμάτωση αλλά και της μετανάστευσης. Ερωτώ λοιπόν. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο δράσης πώς θα εξασφαλίσουν ότι οι παρανομοί μετανάστες δεν θα χάνονται από τις αρχές μετά την άφηξή τους στην Ευρώπη. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι ΜΚΟ δεν θα καταλήγουν να μεταφέρουν σε ευρωπαϊκή επικράτεια ε, ενδυνάμει τρομοκράτες. Ε, και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ισλαμική προπαγάνδα online και μέσω των μάμιδων θα ανακόπτεται εγκαίρως για να σώζονται ζωές και να μην ε, ενισχύονται τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Ευχαριστώ πολύ.

Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt. Jetzt, hören Sie. Sehr gut. Με ακούτε? Πολύ ωραία. Κυρία Επιτροπέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Νομίζω ότι μετά από τις τρομακτικές επιθέσεις βλέπουμε συνέχεια να επαναλαμβάνονται τα ίδια συναισθήματα. Ακολουθούν νέες προτάσεις, προτάσεις οι οποίες περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το ζήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω λοιπόν να σας ρωτήσω με σαφήνεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύει για τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για περιορισμό των ε, ελευθεριών. Θα υποβάλει σχετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε. Και Επίσης θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση σε ό,τι αφορά την τήρηση και αρχιοθέτηση των δεδομένων. Ευχαριστώ. Ε, Jorge Busade, conectado. Ναι, ευχαριστώ, λέει ο Μπουσαντέ. Μιλάμε μια στρατηγική αντιμετώπιση τη τρομοκρατία. Όμω, ε, όπω είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, διαπιστώνουμε ότι πρέπει να πάμε στο βάθος των πραγμάτων, να έχουμε μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση. Βεβαίως ε, και οι τρεις καθολικοί που δολοφονήθηκαν στην Νίκαια, ε, του σκότωσε ένας ε, τρομοκράτης, παράνομος μετανάστης που από την Απεντούσα. Ο, ο, η δολοφονία του καθηγητή στη Γαλλία ήταν ένας ψευτοπρόσφυγας που τον σκότωσε. Βεβαίω μπορούμε να κατηγορήσουμε του Ευρωπαίου ή να κατηγορήσουμε και τον καθηγητή. Ε, ο οποίος ασκούσε την ελευθερία ε, έκφρασης. Ε, μπορείτε να κατηγορήσετε και εμένα αν νιώσετε καλύτερα. Αλλά πρέπει να έχουμε και μια στρατηγική για να κλείσουν αυτές οι βαχαμπιστικές και οι σαλαφιστικές τα τζαμιά αυτά. Στο νέο σχέδιο λοιπόν για το άσυλο και τη μετανάστευση λείπουν συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει να μπορούμε να στέλνουμε πίσω τους ανθρώπους αυτούς στις τρίτες χώρες. Ε, και οι τρίτες χώρες που δεν συνεργάζονται μαζί μας για την ε, θελούσια επιστροφή ε, θα πρέπει να τιμωρούνται. Δεν είναι... Δεν μιλάμε πλέον για να... Ε, ένα δούριο ύπο που έχει δεν πρέπει να μπει στην Ευρώπη. Έχει ήδη μπει, είναι εδώ οι άνθρωποι αυτοί. Ε, και πρέπει να προστατεύσουμε του συμπολίτες, μα, του μας, μα. Μάλιστα, ωραία, πολλά ακούστηκαν και πολύ έτσι ζωντανά, ζωντανή συζήτηση. Βεβαίω, οι τελευταίε εξελίξει, ε, οι τελευταίε επιθέσει και στη Γαλλία και στην Αυστρία είναι τραγικέ. Ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία που υπάρχει. Και αυτό φάνηκε και στη συζήτηση τα δικαιώματα των θυμάτων, η προστασία των πολιτών, η ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ε, κομμάτια του παζλ, θα προσπαθήσει να τα συνδέσει. Έχουμε λοιπόν πολύ τροφή προσκέψη. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους δύο προσκεκλημένους, ε, την κυρία Γιώχανσον. Κυρία Γιώχανσον πρώτα λοιπόν, αν μπορείτε να μιλήσετε 6 λεπτά αντί για 10 ε, για να μείνουν 3-4 λεπτά και για τον κύριο Κλώσ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω. Ήταν πολλά τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται πιο σύντομα η ασφάλεια επιγραμμικά είναι μεγάλη, μεγάλη προτεραιότητά μου. Ορισμένε φορέ έχω την εντύπωση ότι είμαστε αγαθοί. Πρέπει να προστατεύουμε, να προστατεύουμε καλύτερα στο διαδίκτυο. Βεβαίω πρέπει να προστατεύουμε το, την ελευθερία του λόγου, αλλά να, πρέπει να προστατεύσουμε όπω ο Σαμιέλ Πατή, ο καθηγητή, ο οποίο ήταν υπέρ τη ελευθερία του λόγου και τον σκότωσε ένα τρομοκρατή που που τον βρήκε στο διαδίκτυο. Ε, πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε, να προλάβουμε ε, και να απαντήσουμε σε αυτές τις επιθέσεις. Πολλοί είπαν ότι οι τρομοκράτες θέλουν να καταστρέψουν την κοινωνία μας και επιτίθεται στις αξίες μας και χρησιμοποιούν την ελευθερία που υπάρχει στο διαδίκτυο γι' αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι. Το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν τώρα είναι ήδη υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνονται εκεί ε, στοιχεία που έχουν να κάνουν με τρομοκρατία. Όμως όλοι όσοι μπαίνουν στη Σέγγεν δεν, δεν περνάνε από το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν όπως λέει η Frontex και αυτό με ανησυχεί. Βεβαίως κάποιοι τρομοκράτες έρχονται εδώ, περνάνε τα σύνορα με τον στόχο να διαπράξουν κάποια κλιματική πράξη, κάποια τρομοκρατική πράξη. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να προστατεύουμε του συμπολίτε μα, γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε. Και γι' αυτό λέω πρέπει να υπάρχει μια υποχρεωτική διαδικασία screening για όποιον μπαίνει παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει αυτόν να εισάγεται στο, πρόγραμμα, στο σύστημα Eurodac και αν αποτελεί απειλή να μην του επιτρέπεται να εισέλθει στο έδαφο τη Ένωση. Όμω η μετανάστευση είναι κάτι φυσιολογικό Έχουμε 22 εκατομμύρια ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προέρχονται από τη μετανάστευση. Και δεν έχουμε βεβαίω 22 εκατομμύρια ανθρώπου που μα απειλούν. Είδαμε τον νεαρό Παλαιστίνιο, ο οποίο έσωσε ε, αστυνομικού στην προηγούμενη επίθεση. Σε ό,τι αφορά ε, τώρα την απόφαση του Πριμ και την. Ε, οδηγία API ε θα τα παρουσιάσουμε αυτά στην αρχή του έτους. Τώρα για τον ε, ορισμό του τρομοκράτη. Αυτά είναι σαφές στον κανονισμό. Ε, χρειάζεται συνεργασία. πρέπει να είναι η συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών θα πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η αναπερίπτωση. Η API και το PRIM δεν έχουν να κάνουν με τη συλλογή νέων δεδομένων. Θέλουμε να έχουμε πιο σύγχρονους τρόπους ανταλλαγής των δεδομένων για το πριν παραδείγματο χάρη θέλουμε να έχουμε ένα κεντρικό router να υπάρχει μία σύνδεση από τα κράτη-μέλη ε, σε ό,τι αφορά την, τον, τον, τον, ε, την διάχυση την, το να μοιραζόμαστε τα hit με άλλες χώρες το API τώρα έχει να κάνει με την καλύτερη ποιότητα των δεδομένων που ήδη στέλνουμε ε, στα κράτη-μέλη που μας το ζητούν. Να είναι πιο ποιοτικά τα στοιχεία αυτά και να είναι πιο επικαιροποιημένα. Και να υπάρχει μια πιο σύγχρονος τρόπος προστασίας των δεδομένων αυτών. Πρέπει να πω ότι βλέπω ότι το PNR ε, αναφέρθηκε, αλλά δεν προετοιμάζουμε κάποια αλλαγή από αυτού. Έγινε συζήτηση για την κρυπτογράφηση. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό, βεβαίω. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την κυβερνοασφάλεια για την προστασία των δικαιωμάτων, όπω η ιδιωτική ζωή. Ταυτόχρονα, η κρυπτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από του ίδιου του εγκληματίε για να αποκρύψουν τι πράξει του από τι αρχέ επιβολή του νόμου ε, και θα είναι δύσκολο να τους εντοπίσουμε και να τους διώξουμε. Ε, Γι' αυτό λοιπόν λέμε στην στρατηγική για την ασφάλεια της Ένωσης που θα παρουσιάσουμε το Δεκέμβρη ότι θα πρέπει να βρούμε ισορροπημένες λύσεις τεχνικές, νομικές ε, για την κρυπτογράφηση προστατεύοντας την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των επικοινωνιών αλλά ε, να είναι ταυτόχρονα και εργαλεία αποτελεσματικά, αποδοτικά για τις αρχές υποβολής του νόμου. Ως ε, πολιτικοί θύνοντες πρέπει να βρούμε το κατάλληλο σημείο ισορροπίας εδώ οι τρομοκράτες αποτελούν απειλή και θα πρέπει να προστατευτούμε πολύ καλύτερα και σε ό,τι αφορά τη στρατολόγηση των ανθρώπων αυτών που και αυτή γίνεται στο διαδίκτυο σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν αυτές οι κοινότητες μίσους όπου εμπνέουν οι μεν τους δε, μαθαίνουν οι μεν τους δε ε, πώς να ριζοσπαστικοποιηθούν. Πρέπει λοιπόν το περιεχόμενο το τρομοκρατικό που ε, εντοπίσουμε στο διαδίκτυο να κατεβαίνει αμέσως. Πρέπει να υπάρχει μια εθνική αρχή αρμόδια ε, που θα αποσύρει οποιοδήποτε τέτοιο υλικό και διασυνοριακά να διαχέει πληροφορία αυτά ε, στα άλλα κράτη-μέλη και να μπορεί να διωχθεί οποίο έχει ανεβάσει το περιεχόμενο αυτό. Αλλά το πιο βασικό είναι να κατέβει αμέσω το περιεχόμενο. Τώρα για τη Σέγγεν. Προετοιμάζουμε το πρώτο φόρουμ για το Σέγγεν που θα λάβει η χώρα σε μερικέ εβδομάδε. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση για το μέλλον του Σέγγεν και τι εξελίξει που ε, θα είναι απαραίτητε. Θα τα παρουσιάσουμε αυτά στη στρατηγική μα για τη Σέγγεν το Μάιο του χρόνου. Δεν θέλουμε εδώ να προσθέσουμε νέα στοιχεία, νέε πληροφορίε. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις υπάρχουσες πληροφορίες, με καλύτερη διασύνδεση, με καλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων ε, συστημάτων. Το σχέδιο δράση τώρα για την ένταξη και την ε, ενσωμάτωση θα το παρουσιάσουμε τον ερχόμενο μήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις ΜΚΟ στο τοπικό επίπεδο, διότι εκεί λαμβάνει η χώρα η ένταξη, εκεί λαμβάνει η χώρα η ενσωμάτωση και εκεί μπορεί κάποιο ε, να ε, βρει, ε, έχουν φίλους, να κάνει φίλους, να βρει γνωστούς. Είναι πολύ, παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο δηλαδή αυτοί οι παράγοντες και οι τοπικές αρχές ε, στην ένταξη και την ενσωμάτωση. Για την καλύτερη προστασία των συνόρων είναι απαραίτητη προφανώς Τώρα για την πρόληψη. Και η πρόληψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν είμαστε καλοί στην πρόληψη, όταν τα καταφέρνουμε σε επίπεδο πρόληψης, τότε ε, μπορούμε ε, να σταματήσουμε τη ρεσπαστικοποίηση. Βέβαια, ποτέ δεν θα υπάρχουν πηχαίοι τίτλοι για αυτό, για την πρόληψη, αλλά έχει, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η οδηγία η αντιτρομοκρατική δεν έχει μεταφερθεί σωστά σε όλα τα κράτη-μέλη. Όμως ο ορισμός τρομοκρατίας υπάρχει. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο σε επίπεδο εφαρμογής. Τώρα για το PNR και τη συμφωνία με τον Καναδά. Υπήρξε αντικείμενο σε αυτή η συμφωνία όμως ε, δεν συμφωνούν με σε ό,τι αφορά το κείμενο. Το τελικό για την ώρα έχει λογαριστεί διαπραγματεύσει τώρα για το Brexit. Είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε μια καλή συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφάλειας. Όμως αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι η κατάλληλη συγκυρία για να πούμε τι θα γίνει αν δεν φτάσουμε σε συμφωνία. Διότι βρισκόμαστε ακριβώς ε, το πιο ε, κρίσιμο σημείο της διαπραγμάτευσης. Σας ελπίσουμε ότι θα έχουν θετική έκβαση αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επιτροπέ Γιωχάνσον. Διευκρινίσατε πάρα πολύ τις ερωτήσεις που μας ακούσαμε και κάνοντα το καλύτερο για την ολοκληρώσετε σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Τρία λεπτά. Γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που προβλεπόταν για το θέμα αυτό. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Γερμανικής Προεδρίας για να δούμε κατά πόσο σας βλέπουμε. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρα, και ελπίζω να με βλέπετε καλύτερα τώρα. Έχω τρία λεπτή λεπτά. Να αναφέρω όσο πιο πολλά γίνεται λοιπόν. Η δήλωση. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω γερμανικά. Η δήλωση των Υπουργών Ιστορικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι αρκετά ανοιχτή και η αφορμή ήταν η τρομοκρατική επίθεση, αλλά και ο Ισλαμικός, η ε, Ισλαμική τρομοκρατία, αλλά η διατύπωση περιλαμβάνει και άλλες μορφές τρομοκρατίας, όπως ο δεξής εξτρεμισμός. Έχουμε λοιπόν αυτή την απειλή του εξτρεμισμού της δεξιάς ε. στη Γερμανία. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. οι διάφορες μορφές εξτρεμισμού δεν μπορούν να κλιμακωθούν ανάλογα με την επικίνδυνοτητά τους. Όλες οι μορφές εξτρεμισμού πρέπει να, να καταπολεμηθούν. Θα ήθελα να μιλήσω για το πολιτικό Ισλάμ ως φαινόμενο. Είναι σημαντικό να γίνει και η διάκριση με το θέμα της άσκησης ε, της θρησκείας. Ο πολιτικός Ισλαμισμός είναι κάτι ε, επί του οποίου τοποθετήθηκαν με σαφήνεια οι Υπουργοί Ιστορικών. Είπαν ότι χρειαζόμαστε μέτρα για αυτό το φαινόμενο. Ακούσουμε και κριτική στις δηλώσεις για το κατά πόσον χρειάζονται πραγματικά νέες αρμοδιότητες ή υπηρεσίες ασφάλειας. Υπάρχουν τρεις παράγοντες οι οποίοι αποτελούν, αποτελούν ε, έναυσμα για έρευνα και για την τρομοκρατία και για άλλες, ε, άλλες ε, μορφές εγκλήματος ε, σε θέματα επικοινωνίας και σε σχέση με πρώτερα οδικήματα, εγκλήματα που έχουν διαπραχτεί. Αυτά είναι τα στοιχεία που οδηγούν σε κοινέ βάσεις δεδομένων PI, PNR Μόνο μέσω τέτοιων καταχωρήσεων καταλήγουμε σε διαπίστωση των, του τι συμβαίνει. Ε, επικοινωνία έγινε μέσω όχι πλέον ε, τηλεφώνων. Ο κόσμος πλέον επικοινωνεί μέσω Messenger. Ε, και έτσι λοιπόν το Συμβούλιο δεν καταλήξει σε κάποιο οριστικό συμπέρασμα αλλά σίγουρα θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα αυτό περαιτέρω. Η Επίτροπο δήλωσε και εξήγησε πάρα πολύ καλά γιατί χρειαζόμαστε το πριμ σε ό,τι αφορά ε, τα δακτυλικά αποτυπώματα, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την ε, συλλογή άλλων στοιχείων. Όλα αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν την ε, δικτύωση πληροφοριών, την σύγκριση πληροφοριών και δεδομένων αυτό χρειάζεται από πλευρά ασφάλεια. Και έτσι, σε ό,τι αφορά τους κατηγορούμενους, τους υπόπτου τρομοκρατικών ενεργειών, σε αυτούς ε, απευθύνονται τα μέτρα αυτά, όχι στο ευρύ κοινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, και ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Αυτά λοιπόν την στρατηγική αυτή για την ασφάλεια σε ό,τι αφορά και τις ε, επιθέσεις που πρέπει να δοθούν μετά τις εγκληματικές ε, και τρομοκρατικές επιθέσεις στην Γαλλία και στην Αυστρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, στο σημείο 8, Ευρωπαϊκή Ένωση και η στρατηγική για την Ασφάλεια. Είμαι ο Γιατί εξετάζουμε το σχέδιο ψηφισματο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια και ω συντονιστέ αποφασίσαμε στις 7 Σεπτεμβρίου να προετοιμάσουμε ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό. Είχα την τιμή να το αναλάβω ως εισηγητής. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν το έγγραφο και μετά θα ξεκινήσει ένας γύρος ε, συνομιλίας με τους σκιώδεις εισηγητές. Θα σας παρουσιάσω εν συντομία λοιπόν την έκθεση αυτή. Το σχέδιο λοιπόν κειμένου ε, έρχεται μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2020 για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 έως το 2025. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θεωρεί ότι θα πρέπει να εντοπιστούν το μη προτεραιότητας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει θέματα ασφαλείας. Τέσσερις βασικές προτεραιότητες λοιπόν ορίζονται αντιμετώπιση των απειλών προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από την τρομοκρατία οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ανθρώπων, ε, λάθρεμπορων ναρκωτικών και υποστηρίζοντας ε, το σύστημα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική λοιπόν ε, συνοδεύεται από τρεις βασικές πρωτοβουλίες. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής ε, κακοποίησης παιδιών, ε, σε ό,τι αφορά επίσης ε, το τράφικινγκ, του λαθρεμπόριο όπλων και επίσης βασίζεται σε ήδη υφιστάμενες νομοθεσίες. Η στρατηγική λοιπόν προτείνει νέα στρατηγικά και νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα. Έχουμε λοιπόν μία σειρά νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων. Στο σχέδιο ψηφίσματο, λοιπόν, σχεδιαζόμαστε στην αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις βασικέ. Ε, ε, στα βασικά στοιχεία τη στρατηγική που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει, λοιπόν, να βασιστούμε σε αξίε στο άρθρο 2 της συνθήκη ε, συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει ίση αξία με την ίδια συνθήκη. Ο σημείο κίνηση λοιπόν. Θεωρούμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της ε, εσωτερική ασφάλειας θα πρέπει να υλοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο που τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για την ιστορική ασφάλεια. όπως η Οδηγία 2011-93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δεκεμβρίου του 2011 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και των θυμάτων που δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, δεν έχει υλοποιηθεί από κάποια κρατημέλη. Κατά δεύτερον, τα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα θα πρέπει να ακολουθούν τα κενά που εντοπίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά οποιαδήποτε συγγνώμη, οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να συνδεύεται από μελέτη αντικτύπου. Επιμένουμε από αυτού, γιατί δεν υπάρχει τέτοια μελέτη αντικτύπου σε διάφορες προτάσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς συστηματικά αντιτιθέμεθα όταν δεν υπάρχει αυτή η μελέτη αντικτύπου. επικεντρωνόμαστε σε βασικούς τομείς ε, εγκλήματος, κατάχρηση παιδιών, online, ε, παράνομα ναρκωτικά, ε, τρομοκρατία. Για την τρομοκρατία, ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων το 2009 μειώθηκε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα δυστυχώς αποδεικνύουν το θλιβερό γεγονό ότι υπάρχει ακόμα αυτή η απειλή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η νέα ατζέντα κατά τρομοκρατικών επιθέσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το τρομοκρατικό περιεχόμενο που εντοπίζεται online. Ε, πρέπει να ολοκληρωθεί το θέμα αυτό. Εργαζόμαστε από αυτό με συνδυασμό νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων. Για την καταπολέμηση λοιπόν της τρομοκρατίας έχουμε επαναλάβει και έχουμε ζητήσει την αναθεώρηση του, σε αποφασής πλαισίου του Συμβουλίου του 2008 για να υπάρχει καταρχάς ένας κοινωνός ορισμός για το οργανωμένο έγκλημα και για την υλοποίηση της ε, αποφασής πλαισίου. Για την αποτελεσματική λοιπόν καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Έχουμε την σεξουαλική κακοποίηση online. Εδώ υπάρχει εντατική και επίγουσα ανάγκη να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε ε, μορφή σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών online και offline. Και επίσης να καταπολεμήσουμε το περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης online. Θα συνεχίσουμε ε, να εργαζόμαστε με την ε, αποκλήση e-privacy την οποία έχουμε την πραγματική την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε το θέμα λοιπόν τη σεξουαλική κακοποίηση online και περιμένουμε σχετική ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τα ναρκωτικά για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να προστατεύσουν του πολίτε ε, από τι απειλέ που συνδέονται με τα ναρκωτικά. Η ευρωπαϊκή λοιπόν πολιτική για τα ναρκωτικά θα πρέπει να συνεχίζει να ενσωματώνεται βάσει μιας ε, ε, πολυτομιακής προσέγγισης. Τέλος, η σημασία της ευρωπαϊκής ασφάλειας σε ό,τι αφορά τις θεσμικές ρυθμίσεις, η Γυροπόλης, οι η Γυροτζάστα αποτελούν πυλώνας του συστήματος αυτού ε, οργανώσεων που καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους. Η αναθεώρηση της εντολής της Γυροπόλ και ο Κανονισμό για την προστασία δεδομένων του GDPR. Αλλά και ο κανονισμός του 2017. Το DPS θα αναθεωρηθεί για τη βάση δεδομένων που διατηρείται στη Europol σε ό,τι αφορά το μελλοντικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο. Όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν με τη δουλειά που κάνουμε προκειμένου να υπάρχει αυτό το σύστημα διαλειτουργικότητας το οποίο επιθυμούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα. Έχουμε και τους περιορισμούς της μετάφρασης και του καθεξής. Αυτά είναι οι περιορισμοί της δουλειάς μας. Προσπαθούμε λοιπόν να ενσωματώσουμε την δουλειά των πολιτικών ομάδων σε όλο το οικοδόμημα το οποίο έχουμε μπροστά μας, αλλά υπολογίζω και στη δική σας σύμβολη. Περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας, θέλετε συνεργασία σας, για να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι συνεκτικό, θα ορίζει τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της ε, εσωτερικής ασφάλειας για τα επόμενα 5 χρόνια, 2020 μέχρι 2025. Ας, Ας ακούσουμε λοιπόν τους ε, ισχυοδησίτες πρώτους, του κ. Αλέχος. ¿Estás ahí? Nope. Ο κύριος Σαρθαλέχος. Ναι, παρακαλώ, ναι. Ελπίζω τώρα να με ακούτε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ και ως εισηγητή για το έργο σου ε, και για το έργο που ετοιμάζεσαι βεβαίω να συνεχίσει να κάνει. Ε, αυτό το σχέδιο ψηφίσματο εμεί το εξετάζουμε σε μια στιγμή όπου όχι μόνο βρισκόμαστε ε, εν μέσω πανδημίας αλλά έχουμε και την επανεμφάνιση της τρομοκρατικής απειλής. Η πραγματικότητα λοιπόν μας δείχνει ότι η κρίση ασφάλειας δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι κάτι το οποίο θα το βρίσκουμε συχνά, μας, συχνά μπροστά μας. Και αυτό ε, θα έρχεται να δοκιμάσει όχι μόνο τις, ε, την δύναμη, την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών μας, αλλά και τη δυνατότητα διαχείρισης των κρίσεων αυτών από την πλευρά μας. Διαπιστώνουμε ότι το σχέδιο ψηφίσματος ε, είναι ε, καλό, το βλέπουμε θετικά, ξέρουμε ότι ήταν δύσκολες οι συνθήκες εκπόνησής του. Ε, Βεβαίω η τρομοκρατική απειλή όπως εμφανίζεται τη στιγμή παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο διότι η τρομοκρατία αυτή τη στιγμή ε, αλλάζει, μεταλλάσσεται και πέρα από τα κλασικά προβλήματα τρομοκρατίας που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση υπάρχει ένα πρόβλημα ριζοπαστικοποίησης. Ριζοπαστικοποίηση στις φυλακές, ριζοπαστικοποίησης μέσα στην κοινωνία. Είναι απαραίτητο αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Ε, καθώς και το θέμα του ελέγχου στα σύνορα. Δεν λέω εγώ πόσοι πρέπει να μπουν στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει από πλευρά ασφάλεια είναι ποιοι είναι αυτοί, όχι πόσοι. Και εδώ χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, έχει γίνει σχετική αναφορά, για τα δεδομένα, για τα μέσα που θα μα επιτρέψουν να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για αυτού του ανθρώπου. Χρειαζόμαστε λοιπόν στρατηγικέ κατά τη Ε, υπάρχουν ήδη κάποιε, πρέπει να τι βελτιώσουμε και να τι ενισχύσουμε. Είναι σημαντικό επίσης να δώσουμε έμφαση στην αναγκαιότητα δικαστικής συνεργασίας. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα, ε, ένα χώρο ελευθερίας και ασφάλειας κοινό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ιδίως εάν θέλουμε αυτός ο χώρος ε, ασφάλειας ε, να μην οικοδομηθεί σε βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σημερίζομαι με τον εισηγητή την άποψη ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων. Είναι οι αριθμοί πραγματικά αποστομωτικοί, τα έχουμε ακούσει ξανά και ξανά και η διαφοροποίηση μεταξύ online και offline ε, κάποια στιγμή πάβει να υπάρχει και πολύ συχνά η παρενόχληση αλλά και η σεξουαλική κακοποίηση επιγραμμικά είναι ένα, ε, μια πρώτη φάση πριν την πραγματική σωματική κακοποίηση. Ε, επίσης θέλω να πω ότι η Europol είναι ένα σημαντικό όπλο ε, στο σύστημά μας και θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την εντολή της Europol. Τέλος, ε, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο και στην Επιτροπή αυτή ότι η τεχνολογική πρόοδος ε, δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε διότι η ασφάλειά μας θα έχει ένα, μια τεχνολογική διάσταση όλο και πιο σημαντική, μια ψηφιακή διάσταση και αυτό βεβαίως ε, θέτει νέα ζητήματα που έχουν να κάνουν και πάλι με την διαφύλαξη των θεμελιών δικαιωμάτων και τις βασικές αξίες, τι βασικέ αρχέ μας σε νομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό το σχεδίο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας ε, που θα μας επιτρέψει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης να έχουμε κοινέ πολιτικέ, κοινέ στρατηγικέ, Δεν αρκούν μόνο νομοθετικά πλαίσια, πρέπει να ενισχύσουμε συγκεκριμένες στρατηγικές που περνούν από τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα Θαρθαλέχος. Οι υπόλοιποι παρακαλώ σεβαστείτε το χρονικό όριο. Ε, βεβαίως και σημειώνω όλα τα σχόλιά σας, αλλά παρακαλώ ως συνήθω έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε μέχρι τις 7 παρατέταρτο, άντε μέχρι τις 7 παρα 10 το πολύ. Μετά θα πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Ε, και έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε σημαντικά, όπως ε, η εξαίρεση που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τις επικοινωνίες σε σχέση, με το e-privacy οπότε παρακαλώ να είστε όσο γίνεται πιο συνεκτικοί στις παρεμβάσεις σας. Τον λόγο έχει τώρα ο, ο Ντράγκος του Ντουράτσε από τη Ρινιού. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, ο κύριος Τοντοράτσε. Uh, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Συμφωνώ με πολλά από τα όσα έχεις εδώ αναφέρει συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου ε, για τις, ε, ε, από τις νέες αυτές προτάσεις. Θέλω να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την ψηφιοποίηση. Η στρατηγική αυτή είναι ελπίσω όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία που μπορεί να διευκολύνει την καταπολέμηση του εγκλήματος αλλά και μπορεί να διευκολύνει το ίδιο το έγκλημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένες ε, λύσεις και θα κάνω κάποιες ε, τροπολογίες. Τώρα, ε, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και συνδυάζεται με τα όσα είχατε πει και εσείς για την Europol, ότι δηλαδή θα πρέπει να ενισχύσουμε την εντολή της Europol, το χρειαζόμαστε αυτό, αλλά... Υπάρχει μια σημαντική απουσία σε το πλαίσιο της στρατηγικής που είναι το VPPO. Δεν υπάρχει τίποτα για το VPPO στην στρατηγική, ενώ υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην διαφθορά και τα οργανωμένα εγκληματικά συνδικάτα τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω της χρήσης project που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά χρήματα. Και κάπως πρέπει αυτό να το αναχαιτήσουμε μέσω της στρατηγικής της Ένωσης. Αυτό λείπει λοιπόν από τη στρατηγική μας και χρειάζεται πιστεύω στο ψήφισμα κάτι να πούμε σχετικά. Άλλη παρατήρηση σχετίζεται με το ρόλο της εκπαίδευσης όσον αφορά την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Θα δεν υπάρχει βάση στη συνθήκη όσον αφορά την εναρμόνιση των, της ύλης όσον αφορά την εκπαίδευση, αλλά Πιστεύω πως είναι σαφές ότι εφόσον θέλουμε να καταπολεμήσουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την ριζοσπαστικοποίηση, θα πρέπει να εστιάσουμε στην παιδεία, να εστιάσουμε στο θέμα της, του φύλου, της ισότητας, ε, για να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας τέταρτη παρατήρηση που θέλω να κάνω συνδέεται με μια επίσης σημαντική απουσία από το κείμενο αυτό που αφορά τις ψευδείς, τα ψευδή νέα και την παραπληροφόρηση. Δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου αυτό το θέμα στο κείμενο, ενώ πιστεύω πως είναι θέμα ασφάλειας για την Ένωση και ε, θα προβώ σε συγκεκριμένες προτάσεις ε, για να προσθέσουμε κάποια απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να μείνετε στα δύο λεπτά. Η Σκιώδηση. Σάσια, είστε παρούσα, και Μπρικμά. Μπρικμό. Μάλιστα είμαι εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τη Γραμματεία για το πρώτο σχέδιο. Εδώ θα πρέπει να οργανιστούμε καλύτερα για να αποφύγουμε τις πολύ, τεχνικές, πολύ σύντομες προθεσμίες. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο, είναι θεμελιώδες κείμενο, πολύ σωστό για τα θέματα ασφάλειας δεδομένων των διαφόρων ε, ε, αλλαγών που θέλουμε να δούμε. Οι τελευταίες απόπειρες ε, ε, στην Αυστρία μας δείχνουν πόσο η καταπολέμηση των δογμάτων ε, παραμένει με μακρύς αγώνας μπροστά μας. Θα πρέπει λοιπόν να θυμίσουμε το κοινωνικό και οικονομικό, κοινωνικό, οικονομικό πλαίσιο το οποίο είναι δύσκολο. Δεν θα πρέπει να, να αποφύγουμε να πέσουμε στις παγίδες, δηλαδή να συγχαίουμε την ασφάλεια με τη διαχείριση των, της μετανάστευσης στα σύνορα. Πρέπει να υπάρχει σωστή διάκριση ανάμεσα στα δύο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να λειτουργήσουμε με βάση τι αξίε μα, ε, το δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το σεβασμό τη ιδιωτική της ιδιωτικής ζωή και τη προσωπική ζωή κτλ. Αναφέρθηκα και από του προηγούμενου να είτε να προχωρήσουμε στο να αξιολογήσουμε τα μέτρα που έχουν προσληφθεί για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του και να γίνουν και μελέτε σκοπιμότητα. Αυτό δεν γίνεται τώρα μέσα στο πλαίσιο τη μεταρρύθμιση του, του καταστατικού τη Europol. Πιστεύω πω πρέπει να τα συνδέσουμε ωστόσο για να αποφύγουμε να μην νομιμοποιήσουμε ε, ε, ε, κάποιες πρακτικές γιατί η, η, η, η πράξη πρέπει να προσαρμοστεί στον νόμο και όχι το αντίθετο. Ε, έπειτα, οργανωμένο έγκλημα το θέμα του ΕΛΚ, ε, πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε σε αυτό το ψήφισμα, η υπενθύμηση του νομικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούμε, αλλά και η ανάγκη ε, για ανθρώπινους και ε, και, και χρηματοπιστωτικούς πόρους. Έχουμε το θέμα της κατάρτισης ε, των ε, δυνάμεων διατήρησης της τάξης, ώστε να, μην, να περιοριστεί και η αστυνομική βία και να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή να δώσουμε στους πιο ευάλωτα, στα πιο, πιο ευάλωτα θύματα ε, τους ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα επιδερμίδας και του, είναι ανάγκη να ενισχύσουμε την πλαισίωση του ελέγχου της συνεργασίας ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό ε, τομέα. Ε, να τονίσουμε τη συνεργασία και με τρίτες χώρες στον τομέα της ασφάλειας. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στις δικές μου τροπολογίες και ευχαριστώ για τη μελλοντική μας συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ναι, βεβαίω έχουμε σημειώσει τη συμβολή σα. Έχετε διαπιστώσει, έχετε τονίσει τη σημασία τη κατάρτιση των αστυνομικών, την προστασία των θυμάτων, ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων. Των... Βεβαίω, όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Δεν έβαλα όλες αυτές τις λεπτομέρειες λόγω ε, μεγέθους. Ε, της έκθεσης, αλλά βεβαίω είναι πολύ σημαντικά και σημαντικό να προσθεθούν μέσω των τροπολογιών, τις οποίες θα περιμένω βεβαίω και σας ευχαριστώ και των προτέρων για αυτές. Επιμένω πάλι στο ε, χρόνο, μείνετε στα δύο λεπτά γιατί έχουμε ακόμα ένα σημείο και τώρα σε λίγο ε, θα, οι διερμηνείς θα διακόψουν. Παρακαλώ. Η κυρία Κάνκο Ασίτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ελευθερία δεν είναι δωρεάν και η ασφάλειά μας δεν είναι δεδομένη. Η Ευρώπη δέχτηκε πάλι επίθεση κατά του τρόπου ζωής της. Και μετά από τις επιθέσεις ε, του Παρισιού πριν από πέντε χρόνια, έπρεπε να δούμε την υπερξιακή απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ο έκτοτε η Ευρώπη ε, στην ουσία εκθρέφει ε, τζιχαντιστές τα κενά στην ευρωπαϊκή ε, ε, πληροφόρηση έχουν επιτρέψει σε πολλούς από αυτούς τους ε, ξένους μαχητές να κινούνται ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα θεμέλια θα πρέπει να είναι ισχυρότερα και βαθύτερα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ατζέντα για, ως ευκαιρία για να ε, καλύψουμε τα κενά που εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες, ε, να μπορέσουμε να πείσουμε τις πλατφόρμες να αφαιρούν το προπαγανδιστικό ε, περιεχόμενο, να έχουμε πιο αποτελεσματική ανταλλαγή στοιχείων και πιο μεγάλες και ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων. Πρέπει να έχουμε πιο διαφανείς κανόνες κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και να μπορούμε να ε, σταματήσουμε τις οργανώσεις που ε, κηρύσουν το μίσος. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεπείς και αποφασιστικές πολιτικές που θα ε, ε, ε, μπορέσουν να καταπολεμήσουν το μίσο στη βία στις κοινωνίες μας. Όσον αφορά την ασφάλειά μας, χρειάζεται μια Ευρώπη που να λειτουργεί και που να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Έτσι θα πρέπει να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τους δεσμούς μας, γιατί για πολύ χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λειτουργήσει εξετάζοντας με μονομένους φακέλους. Αυτό δεν το λέω για να υποβαθμίσω το έργο της αστυνομίας μας και των ε, ε, ε, είμαι ασφαλεία. Αλλά επειδή πρέπει να φτιάξουμε μια πραγματική ένωση με ασφάλεια, ε, πιστεύω πω ω κοινότητα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ισχυρό και φιλόδοξο ε, κείμενο. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Κάνκο. Σημειώσαμε τις πατρίες σας και τώρα περνάμε στην Κορνίλια Ένστ, ε, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι σημαντικό. Να το πω έτσι. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε, αποτελεί ένα πολύ σοβαρό καθήκον. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε διάκριση για το τι ακριβώς μιλάμε, τι εννοούμε ακριβώς και εδώ να πούμε ότι δεν μιλάμε μόνο για Ισλαμική τρομοκρατία. Φυσικά και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο αποκλειστικά για το θέμα αυτό. Το, το είπα και προηγουμένως, έχουμε και άλλο εξτρεμισμό, έχουμε τον εξτρεμισμό των ακροδεξιών. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε όλες τις μορφές της τρομοκρατίας και πώς παρουσιάζεται online, offline. Ξέρουμε επίσης ότι δεν παίζονται όλα στα σύνορα και είναι παράλογο να εστιαστούμε εκεί γιατί η τρομοκρατία γεννιέται στο κεφάλι. Πώς μπορούμε λοιπόν να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, ποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν είναι μόνο η αστυνομία και η εισαγγελία που θα πρέπει να μας βοηθήσουν. Θα πρέπει να θέσουμε τα δύσκολα ερωτήματα. Να δούμε στα κράτη-μέλη τι ελλείψεις υπάρχουν, τι γίνεται με την ισότητα, τι γίνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, με πολλά καυτά θέματα της καθημερινότητάς. Όχι μόνο λοιπόν να εστιαστούμε στα θέματα τη μετανάστευση. Ελπίζω να υπάρξει αυτή η επαναστασία η οποία χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Ένστ και για να γλιτώσουμε χρόνο να πω ότι σημείωσα όλα αυτά που είπατε και προφανώς θα τα ενσωματώσω στην διαδικασία. Σας ευχαριστώ και θα χρειαστώ την συνεργασία σας. Υπολογίζω σε αυτή προκειμένου η τελική έκθεση να είναι όσο πιο ακριβής και όσο πιο συνεκτική γίνεται. Λυπάμαι που περνάμε τόσο γρήγορα στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα, το οποίο είναι και αυτό πολύ επίκαιρο, σε ό,τι αφορά τις προσωρινές αποκλήσεις από την οδηγία e-privacy, ακριβώς για την καταπολέμηση της, κατάχρη... της ε, κακοποίησης των παιδιών ε, στο διαδικτύο. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο πάρα αυτά στην κυρία Σίπελ, για να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Ξέρω ότι δεν είναι απλό. Και πρέπει και εσείς να παρουσιάσετε την ε, υπόθεση αυτή. Σε κάποια λεπτά θα έχουμε μόνο αγγλικά, να το έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω... Για το σημαντικό θέμα όμως, δεν μπορώ σε δύο λεπτά εγώ να το παρουσιάσω. Αντιλαμβάνομαι όλου του περιορισμού, αλλά δεν γίνεται σε ένα τόσο μικροχρονικό διάστημα. Και βεβαίω και οι σκιώδει ηγητέ έχουν το δικαίωμα να και αυτοί να πούν κάτι. Οπότε θα χρειαστώ το χρόνο που προβλέπετε. Θα ήθελα ξεκινώντα να τονίσω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η προστασία των παιδιών σε όλε τι πτυχέ τη ζωή του είναι πολύ μεγάλη σημασία και στο διαδίκτυο και εκτό διαδικτύου. Η εξοργία των παιδιών είναι μια πολύ σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων και αιτιολογεί περιορισμό θεμελιών δικαιωμάτων εφόσον είναι απαραίτητο και αναλογικό αυτό και σέβεται την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Με την έναρξη ισχύ από το Σεπτέμβριο ε, της σχετικής νομοθεσίας το εθελοντικό σκάνινγκ μπορεί να μπει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του ε, e-privacy και θα χρειαστεί οπότε σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων. κάτι που δεν γίνεται. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες που υπάρχουν από το φάκελο αυτό. Υπάρχει και η ανάγκη να υπάρχουν κλίση ασφαλείας στο κείμενο που θα δημιουργούν υποχρεώσεις και για τις εταιρείες αλλά και για τα κράτη-μέλη και ελπίζω το σχέδιο έκθεσής μου να είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να βρεθεί μια καλή λύση το συντομότερο δυνατόν. Να είμαι όμως και σαφής ταυτόχρονα. Βεβαίως και είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και ο φάκελος αυτός. Δεν πρόκειται όμως να υποκύψω σε πιέσεις για να δεχτώ κάτι το οποίο να μην είναι νομικός ε, άτρωτο, να μην μπορεί να το προσβάλλει κανείς θέλω και βεβαίως να είναι προς συμφέρον των παιδιών. Περιπλέκονται τα πράγματα διότι υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου. Η πρόταση υπευλήθη μόλις το Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ο σχετικός κώδικας είχε ήδη αποφασιστεί το Δεκέμβριο του 2018. Χάσαμε σχεδόν δύο χρόνια. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ότι δεν μπορούσε αυτή η νομοθεσία να εγκριθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Υπήρχε μια μικρή πιθανότητα εάν καμία δηλαδή πολιτική ομάδα δεν υπέβαλε τροπολογίες. Όμως εγώ υπέβαλε την πρόταση αυτή στην αρχή της διαδικασίας και δεν έτυχε υποστήριξη, και το καταλαβαίνω αυτό. Διότι ουσιαστικά είναι σαν να ε, παραχωρούμε όλες τις εξουσίες τις κοινοβουλευτικέ. Ταυτόχρονα η Κομισιόν δεν σεβάστηκε την υποχρέωσή τη στα πλαίσια τη καλή νομοθεσία να συνοδεύει την πρότασή τη από μια μελέτη αντικτύπου. Και επιπλέον η Κομισιόν δεν σκοπεύει να πάρει θέση για το κατά πόσο οι εθελοντικέ πρακτικέ που υπάρχουν τώρα για τον εντοπισμό ε, του υλικού κακοποίηση των παιδιών είναι νόμιμα με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κρίσιμε πληροφορίε που έχουν να κάνουν με το επίπεδο ε, διατάραξη των θεμελιών δικαιωμάτων λείπουν έλειπαν κάτι τη στιγμή που προ, προπαρασκευάσαμε την έκθεση αυτή. Αυτό όμω δεν αλλάζει την αποφασιστικότητά μου, τη βούλησή μου να βρεθεί μια λύση όσο γίνεται πιο γρήγορα, εάν μπορούσαμε να τα βρούμε γύρω από κάποιου συμβιβασμού. Εγώ είμαι έτοιμη να πάμε στι 7 και στι 10 Δεκεμβρίου σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Λίμπε. Να σα πω εν συντομία τώρα περί τίνο πρόκειται. Δύο γενικά στοιχεία. Η κρυπτογράφηση από τη μία στην άλλη ε, από την αρχή ως το τέλος είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλίσουμε ε, την προστατευόμενη επικοινωνία και για τα παιδιά και για τα θύματα γενικότερα. Τίποτα λοιπόν στον κανονισμό δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως απαγόρευση ή ως αποδυνάμωση της κρυπτογράφησης από την αρχή ως το τέλος. Επίσης δεν προβλέπουμε, δεν, προβλέπ, δεν συνιστά μάλλον νομική βάση αυτό που προτείνουμε. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, ο κανονισμό πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε βίντεο και σε εικόνε και στην ανταλλαγή ε, mail και μηνυμάτων. Εκεί είναι που η τεχνολογία με βάση τι πληροφορίε που έχουμε είναι εκεί είναι που χρησιμοποιείται περισσότερο. Επειδή λοιπόν έχει προσωρινό χαρακτήρα, αυτό ο κανονισμό πρέπει να είναι περιορισμένο στον παρόν ορισμό σε ό,τι αφορά την παιδική πορνογραφία και την πονογραφική πράξη όπως αυτό αναφέρεται στην οδηγία για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Οπότε φεύγει το grooming, μιας και εδώ δεν συνάδει ο σχετικός ορισμό με το ποινικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα παραδείγματα που άκουσα αφορούσαν ε, φωτογραφίε που χρησιμοποιούν και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν χάσε, το photo DNA και άλλες πληροφορίε. Επίσης, η τεχνολογία πρέπει να είναι ουδέτερη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν τη θέση σε ισχύ του κανονισμού που προτείνει η Κομισιόν, εφόσον δεν πληρεί τι προποθέσει. Ποιε είναι λοιπόν οι προποθέσει και ποιε είναι οι κλίδε ασφαλεία που προσθέτουμε εμεί εδώ. Εφόσον θέλουμε να βασιστούμε στον κανονισμό αυτό, θα πρέπει να πληρούμε προποθέσει όπω μια πρώτερη μελέτη δικτύπου σε ό,τι αφορά προστασία δεδομένων και μια υποχρεωτική διαβούλευση σύμφωνα με το GDPR το άρθρο 61D ή 61E ε, του GDPR είναι μια νομική βάση. Δεν πιστεύω ότι τα ε, θεμητά συμφέροντα είναι ε, επαρκή όταν μιλάμε για επικοινωνία, ιδιαίτερα στην επικοινωνία αυτή εμπλέκονται παιδιά. οι αρχές επιβολής του νόμου δεν μπορούν να λαμβάνουν τις πλευρές αυτές χωρίς πρώτερη εξέταση. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί προσφυγής, ε, ένδικα μέσα και επίσης πολύ σημαντικό να μην υπάρξει καμία παρέμβαση σε οποιαδήποτε επικοινωνία ε, που προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρριτο μεταξύ θυμάτων και ε, δικηγόρων παραδείγματος χάρη. Μια περαιτέρω νομική βάση για τις μεταφορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το GDPR. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τον δημόσιο μητρό πρέπει να δημιουργηθεί για, με τις οργανώσεις που δρούν υπέρ των, του δημοσίου συμφέροντος των παιδιών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίηση των παιδιών και μόνο με αυτού πρέπει να μπορούμε να μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Πρέπει οι, οι πάροχοι να, να μας υποβάλουν εκθέσεις. Έξι μήνε μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού. Έτσι ώστε να έχουμε την πρώτη έκθεση όταν η Επιτροπή θα υποβάλει την πρόταση αυτή για το υποχρεωτικό πια σύστημα. Πριν δώσω το λόγο στους κοινούς συζητητές, θα ήθελα να, ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους για τις συνεισφορές τους έως τώρα και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους ενεπλάκησαν όλο το προσωπικό που με βοήθησε υπό πολύ δύσκολε συνθήκε. Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία να θυμίσω σε όλους ότι όταν εργαζόμαστε πάνω σε πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να υπάρχει επαρκές προσωπικό. Σε εποχή πανδημίας ακόμα περισσότερο. Πρέπει να έχουμε τεχνικές δυνατότητες ε, στις, ε, ε, στη διάθεσή μας επικοινωνία και μέσω διερμηνίας, κάτι που λείπει πολύ συχνά, ακόμα και μετά από τόσους μήνες. Κανείς δεν θέλει να σταματήσει τον εντοπισμό και την, την απόκρυψη του πορνογραφικού υλικού που εμπλέκει παιδιά. Όμως παρότι επήγει πάρα πολύ ο φάκελος αυτός, δεν μπορούμε να σεβαστούμε την προθεσμία του Δεκεμβρίου. Θέλουμε να βρεθεί μια τελική λύση αρχές 2021 και καλό τα μέλη, ε, την Κομισιόν αλλά και τη δίκησή μας να μας δώσουν όλους τους πόρους που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ζήπελ. Και τώρα εμείς πρέπει να σα αφήσουμε, συνεχίσουμε χωρίς διερμηνία. Στα... Περνάμε στους κοιόδη και σας θυμίζω να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Κύριε Σερσαλτέχο, παρακαλώ, πολύ πολύ σύντομα. Χαβιέρα, έχεις το λόγο. What you're doing, we are all under enormous pressure to to meet uh, uh, the deadlines